Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, συνεχίζουμε τις εργασίες μας που ξεκινήσαμε σήμερα το πρωί. Είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα ανταλλαγή απόψε με τον κύριο Ποπόφσκιν και στη συνέχεια με την κυρία Άστον με ευρύτερη σύνθεση και συνεχίζουμε με πολύ αξιότιμους προσκεκλημένους. Έχουμε μαζί μας την κυρία Αρνού, εκτελεστική διευθύντρια της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Άμενας. Σας καλωσορίζουμε στην Επιτροπή μας και τον κύριο Χουι αναπληρωτή διευθυντή του Κοινού Οργανισμού Συνεργασίας στον τομέα των εξοπλισμών. Θα αφιερώσουμε λοιπόν το τμήμα αυτό της συνεδρίασης στο ζήτημα των στρατιωτικών δυνατοτήτων. Θα δούμε ποια είναι τα προγράμματα τα οποία ισχύουν αυτή την περίοδο θα αναφερθούμε επίσης σε ένα πολύ ευχάριστο γεγονός στα πλαίσια της κοινή πολιτικής άμυνας και ασφάλειας. Φέτος το καλοκαίρι, τέλος Ιουλίου, υπεγράφει ανάμεσα στον ΟΚΑΡ και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Άμυνας μία διοικητική συμφωνία και μία συμφωνία για την ανταλλαγή διαβαθμισμένων πληροφοριών, ιδιαίτερα αναμενόμενη συμφωνία αυτή προκειμένου να προωθηθεί και να ενταθεί συνεργασία ανάμεσα στους δύο αυτούς οργανισμούς. Φαντάζομαι ότι οι εκπρόσωποι των δύο αυτών υπηρεσιών θα μας μιλήσουν για τη συμφωνία αυτή και πώ θα τους επιτρέψει πραγματικά να προωθήσουν περισσότερο τα κοινά τους προγράμματα. Το ζήτημα των, του στρατιωτικού δυναμικού και ιδίω το ζήτημα του pooling and sharing, όπως λέμε στα γαλλικά, μας απασχόλησε και κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης των Υπουργών Άμυνας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ακούσαμε σήμερα το πρωί τον κύριο Ποπόφσκι, ο οποίος μας είπε ότι έχει προταθεί ένας κώδικας συμπεριφοράς, ο οποίος θα μας επιτρέψει στο μέλλον να καταφέρουμε να καταγράψουμε ποιες είναι οι πραγματικές ανάγκες στα πλαίσια του pooling and sharing και να απασχολήσει αυτά και τα εθνικά στρατηγικά σχέδια, τα οποία εκπονούνται σε κάθε κράτος μέλος. Και από ό,τι κατάλαβε, οι περισσότεροι Υπουργοί Άμυνας τάχθηκαν υπέρ, σαφώς λέτε υπέρ λοιπόν της πρότασης αυτής. Θα μας πείτε ενδεχομένω και εσείς περισσότερα πράγματα στα πλαίσια του pooling and sharing, της συνδεκμετάλλευσης, της συνένωσης και της κοινή χρήσης. Σίγουρα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το μέσο αυτό για την ε, αμυντική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ξέρω ότι ε, εσείς ε, είστε σε επαφή με τους συναδέλφους σας από το ΝΑΤΟ, από την αρμόδια επιτροπή του ΝΑΤΟ. Επίσης έχουμε εκεί επικεφαλής τον ένα νέο στρατηγό. Θα μπορούσατε ενδεχομένω να μας πείτε ποια είναι η κοινή προσέγγιση που υπάρχει και με το στρατηγό Αμπριγιάλ και να μας ενημερώσετε επίσης τι γίνεται με το pooling and sharing και το smart defense, την ευφυή e έξυπνη άμυνα. Κάτι το οποίο σήμερα εξετάζουν οι υπουργοί στα πλαίσια του ΝΑΤΟ. Ενδεχομένω και για αυτό το ζήτημα θα την ενδιαφέρον να μα ενημερώσετε ποιο κάνει τι στα προγράμματα αυτά, σε αυτέ τι σημαντικέ ε, προθέσει. Ευθύ αμέσω λοιπόν, κυρία Κλωτφόν Σαγνού, σα δίνω το λόγο. Σα ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Όντως, ε, όσα συνήθως είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή για μένα το ότι βρίσκομαι εδώ σήμερα προκειμένου να ενημερώσω για το τι κάνει η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Άμυνας όσον αφορά το ζήτημα των στρατιωτικών δυνατοτήτων. Και με τον κύριο Χουιμπρέχτς που είναι σήμερα μαζί μας μπορούμε όντως να μιλήσουμε περισσότερο για το τι μπορούμε να κάνουμε για την κοινή αυτή συνεργασία που μπορούμε να έχουμε ιδίω μετά την υπογραφή της συμφωνίας ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Άμυνας και τον Κοινό Οργανισμό Συνεργασίας στον τομέα των εξοπλισμών. Και προσβλέπουμε ιδιαίτερα στις δικές σας παρατηρήσεις, στην υποβολή των δικών σας των ιδεών. Και πρέπει να σας πω ότι μας ενθαρρύνει ιδιαίτερα το ενδιαφέρον και η υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Διάβασα το σχέδιο έκθεσης για την ε, ευρωπαϊκή πολιτική άμυνας και ασφάλειας και μας χαροποιεί ιδιαίτερα το ότι υπάρχει τέτοια υποστήριξη στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ξεκινώντας από τη μέθοδο την οποία θα ακολουθήσουμε, αυτή στην οποία αναφέρθηκε ο Πρόεδρος. Όντως σήμερα διεξάγεται μια συνεδρίαση των ε, Υπουργών Άμυνα στα πλαίσια του ΝΑΤΟ, για το ζήτημα λοιπόν του στρατιωτικού δυναμικού, των στρατιωτικών δυνατοτήτων. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να γνωρίζουμε ποιο είναι ο καταμερισμό των αρμοδιοτήτων και ποια διαφορά ανάμεσα στο pooling and sharing και το smart defense. Στην ουσία εξυπηρετούν και τα δύο προγράμματα την ίδια ιδέα, τον ίδιο στόχο. Δηλαδή το να καταφέρουμε να έχουμε ένα υψηλότερο επίπεδο αποτελεσματικότητας στις πολιτικές που ακολουθούμε όσον αφορά τις αμυντικές δυνατότητες είτε πρόκειται για τον ΝΑΤΟ είτε πρόκειται για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως πολύ συχνά λέγεται από τους εκπροσώπους πολλών κρατών μελών, είτε, είτε δραστηριοποιούμεθα στα πλαίσια του ΝΑΤΟ, είτε δραστηριοποιούμεθα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν πολλά κράτη-μέλη τα οποία προφανώς συμμετέχουν και στους δύο φορείς, μολονότι η σύνθεση δεν είναι πάντα ίδια, ούτε η μέθοδος εργασίας. Υπάρχει πάντως μια κοινή ομάδα κρατών η οποία παραμένει ίδια και στις δύο φορείς. Κοινός λοιπόν στόχος, αλλά καλύτερη αποτελεσματικότητα μέσω μιας βελτιωμένης συνεργασίας. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως το γνωρίζετε, ελήφθη μια απόφαση από το Συμβούλιο στην άτυπη μάλλον συνεδρίαση των ε, Υπουργών Άμυνας το Νοέμβριο πριν από δύο χρόνια να προωθηθεί η πρωτοβουλία αυτή προκειμένου να έχουμε το περίφημο αυτό pooling and sharing ως μέθοδο, αυτή την συνένωση και κοινή χρήση των στρατιωτικών δυνατοτήτων. Και ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ λίγο αργότερα αναφέρθηκε στην έννοια της ευφυούς άμυνας, smart defense. Για να λειτουργήσουν τα δύο προγράμματα χρειάζεται μια απόλυτα στενή συνεργασία και όπως είπε ο Πρόεδρος με τη συνεργασία του στρατηγού Αμπριγιάρ και όχι μόνο με τον ίδιο. Άλλωστε δεν είναι δύσκολο να υπάρχει μια πολύ καλή επαφή σε τόσο υψηλό βαθμό επίπεδο. Σε όλα μάλλον τα επίπεδα καταφέραμε να πετύχουμε την καλύτερη δυνατή συνεργασία ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Άμυνας, το ACT, έγινε μια πολύ σημαντική εργασία. Περάσαμε σε πάρα πολλές λεπτομέρειες και θελήσαμε να δούμε ποιες είναι οι ανάγκες των κρατών μελών που συμμετέχουν στο ΝΑΤΟ σε ποιους τομείς ε, θέλησαν να δραστηριοποιηθούν όσον αφορά τη μεταξύ ημών συνεργασία και ξεκινώντας από κάποιες πολιτικές προσδοκίες των κρατών μελών προσπαθήσαμε να συνεργαστούμε όσο το δυνατόν καλύτερα για να αποφύγουμε επικαλύψεις και τουλάχιστον στον ιατρικό τομέα αποφασίστηκε από τα κράτη-μέλη τόσο στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και στα πλαίσια του ΝΑΤΟ να υπάρχει μία συνένωση και κοινή χρήση δυνατοτήτων. Αυτό άλλωστε έκανε και η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω ενό προγράμματο κινητών ιατρικών μονάδων στην Ήπεθρο. Και αντίστοιχα προγράμματα έχουν εφαρμοστεί στο Αφγανιστάν. Προσπαθήσαμε πάντως να έχουμε και στις δύο πλευρές, ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση, τα ίδια κριτήρια. Ακόμα και όταν εμπλεκόντουσαν κράτη-μέλη, τα ίδια κράτη-μέλη και στις δύο πλευρές, ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση, προσπαθήσαμε να ακολουθήσουμε μία κοινή γραμμή, να υπάρχει μια κοινή οριοθέτηση των στόχων και να καταφέρουμε με στονισμένο τρόπο να αλληλοσυμπληρώνεται η δράση μας αποφεύγοντας α, τις επικαλύψεις. Ο στρατηγός Παλωμερό την προηγούμενη εβδομάδα μαζί με την συνεδρίαση των Υπουργών στην Λευκοσία μας μίλησε για τα ζητήματα τα οποία έφυξε ο Πρόεδρος, ατύπως μίλησα μαζί του και αυτή τη στιγμή αναλάβει επισήμω τι νέε του αρμοδιότητε, θα ξεκινήσει η επίσημη θεσμική συνεργασία και μαζί του, καθότι όπω είπατε και εσεί, Πρόεδρε, θα είναι επικεφαλή του ACT. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει ο ίδιο συντονισμό δηλαδή και με τι επιμέρου υφιστάμενε ομάδε. Μετά από την σύνοδο του Σικάγο, πολλές από τις δραστηριότητες αυτές θα αρχίσουν να απασχολούν τις διάφορες επιτροπές του ΝΑΤΟ. Πρέπει λοιπόν και το ΝΑΤΟ να καταφέρει να έχει το ίδιο επίπεδο διαφάνειας και συντονισμού σε όλες αυτές τις δραστηριότητες, τις νέες, αφού περάσουν βέβαια στην καθημερινή πλέον εργασία του ΝΑΤΟ. Πιστεύω ότι, θα βασιστούμε και εκεί πέρα και εκεί στην πολύ καλή συνεργασία που υπάρχει ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Άμυνας και το ACT. Οι στόχοι, όπω είπαμε, είναι οι ίδιοι. Υπάρχει μια πολύ καλή συνεργασία. Στι δύο όμω πλευρέ, έχουμε πολλέ φορέ ε, διαφορετικά στοιχεία, διαφορετικά μέσα για να καταφέρουμε να φτάσουμε στο ίδιο αποτέλεσμα. Όσον αφορά το ΝΑΤΟ, είναι σαφές ότι εκεί εποφελούμαστε από το σύνολο των συμμάχων, από όλα αυτά που μπορούν να γίνουν και με τις ΗΠΑ και με τον Καναδά ιδιαίτερος. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για πολλές από τις στρατιωτικές δυνατότητες, στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε άλλου είδους συνέργειες. Συνέργειες με τις άλλες πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συνέργειες με τις ε, δραστηριότητες τις οποίες προωθείτε και εσείς, τις δραστηριότητες αυτές της ασφάλειας που δεν είναι ούτε καθαρά στρατιωτικές ούτε καθαρά πολιτικές. Νομίζω ότι και αυτές θα μπορούσαν να ενταχθούν στα πλαίσια του pooling and sharing. Στη συνέχεια έχουμε όλο αυτόν τον τομέα που συνδέει τις, το στρατιωτικό δυναμικό με, από, με αυτό το οποίο ονομάζουμε στα αγγλικά airworthiness, τον υπάρχει δηλαδή μία συνεκτικότητα ανάμεσα στους κανονισμούς που υφίστανται στον πολιτικό τομέα και στους κανονισμούς που υφίστανται στο στρατιωτικό τομέα και είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορούν οι ίδιοι κανόνες να εφαρμοστούν σε, στα remote piloted systems, στα αεροσκάφη χωρίς κυριστές, στα μη επανδρομένα αεροσκάφη. Και κάτι ακόμα το οποίο θα ήθελα να αναφέρω και το οποίο ουσιαστικά μας εμπλέκει στα πλαίσια, τα task, στα πλαίσια της Task Force της Επιτροπής έχει να κάνει με την έρευνα, την ανάπτυξη, την αγορά και την αμυντική βιομηχανία. Να προσπαθήσουμε δηλαδή και στον τομέα αυτό να καταφέρουμε να καταλήξουμε σε κάποιες κοινέ στρατικές δυνατότητες από κοινού. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Άμυνας θέλει επίσης να εργάζεται και στην βάση της τεχνολογίας που υφίσταται για την άμυνα. Δεν θα πρέπει λοιπόν να ξεχνάμε την διασύνδεση αυτή που υπάρχει με την τεχνολογία και τη βιομηχανική βάση. Να γνωρίζουμε δηλαδή ποιες είναι οι βιομηχανικές δυνατότητες Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της άμυνας και ποιος είναι ο εξοπλισμός ή οι υπηρεσίες που ενδεχομένως να έχουν ανάγκη οι στρατικές μας δυνάμεις. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν να υπάρχει διασύνδεση αυτή και είναι πολύ σημαντικό να καταφέρουμε να υποστηρίξουμε στον τομέα αυτό τα κράτη-μέλη. Ας μην ξεχνάμε ότι η αμυντική βιομηχανία συνεισφέρει στην απασχόληση, στην κοινοτομία και την έρευνα σε όλα τα κράτη-μέλη. Ένα άλλο στοιχείο το οποίο θα ήθελα τώρα να τονίσω είναι ότι το pooling and sharing πρέπει να είναι μια ρεαλιστική μέθοδος εργασίας. Δηλαδή, προσπαθήσαμε να προτείνουμε στα κράτη-μέλη μία μέθοδο εργασία στην οποία θα μπορούσαν ουσιαστικά να προσχωρήσουν, δράσεις τις οποίες θα μπορούσαν να επιτελέσουν. Λαμβάνοντας υπόψη βέβαια και το πολύ ευαίσθητο ζήτημα της εθνικής κυριαρχίας. Και προσπαθήσαμε να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα αυτό σημείο προς σημείο. Τα κράτη μάλι θέλουν να είναι διαθέσιμο το στρατικό δυναμικό εφόσον, εφόσον υπάρχει από την άλλη δεν επιθυμούν να υπάρχει ένα σύστημα απόλυτο αυτοματισμού. Στα πλαίσια ενό συστήματο συνεργασίας θέλουν να ξέρουν ότι υπάρχει μια ασφάλεια εφοδιασμού και ότι τελικά δεν θα υπάρξει κάποιος εταίρο στην όλη αυτή η αλυσίδα που δεν θα ανταποκριθεί στις υποχρεώσει του. Επομένως, θελήσαμε να δούμε πώς θα καταφέρουμε να εμπλέξουμε με τον πιο ρεαλιστικό, ρεαλιστικό με τρόπο τα κράτη-μέλη, προκειμένου να καταφέρουν τελικά να συνεισφέρουν στο στρατιωτικό δυναμικό, χωρίς να προβλέπεται ένα απόλυτα αυτοματοποιημένο σύστημα. Θελήσαμε δηλαδή μία μέθοδο εργασία που θα σέβεται το σύστημα συνεργασία στο οποίο υπάρχει ανάμεσα στα κράτη-μέλη και ιδίω όσον αφορά το ζήτημα του εφοδιασμού. Δεν ξέρω πόσο χρόνο έχω στη διάθεσή μου. Πρέπει να αποχωρήσω στις 3.30. Θα ήθελα τώρα να αφαιρθώ σε τρία σημεία. Πρωτού πάρει το λόγο και ο συνάδελφος από, την, από το Κοινό Οργανισμό Συνεργασίας στον τομέα των εξοπλισμών. Πρέπει καταρχάς να εγκρίνουμε αυτή τη μέθοδο συνεργασίας όσον αφορά τη συνένωση και την κοινή χρήση για συγκεκριμένες στρατιωτικές δυνατότητες. Μόνο κατά αυτόν τον τρόπο θα καταφέρουμε να εξασφαλίσουμε μια αξιοπιστία και θα καταφέρουμε τελικά να εμπλέξουμε όλους τους παράγοντες στον τομέα της άμυνας στα πλαίσια αυτής της συνεκμετάλλευσης. Θέλουμε λοιπόν συγκεκριμένα σχέδια, συγκεκριμένα προγράμματα. Μπορούμε για παράδειγμα να αναφερθούμε στον ανεφοδιασμό, τον εφοδιασμό καυσίμου, Ξέρετε ότι το ζήτημα αυτό μας απασχόλησε και κατά τη διάρκεια της εκστρατείας στη Λιβύη. Οι Ηνωμένε Πολιτείε μας είπαν ότι δεν θα πρέπει να βασιζόμαστε μόνο σε αυτούς, ότι θα αναλαμβάνουν δηλαδή μόνο οι Αμερικάνοι τον ενέργειο εφοδιασμό καυσίμων. Είπαν επίσης ε, ότι ε, μάλλον και το ίδιο θα πρέπει να ισχύει και για άλλες ε, αποστολές όσον αφορά την έρευνα, τον εντοπισμό και την επιτήρηση μας είπαν οι Αμερικανοί ότι θέλουν και εμείς οι Ευρωπαίοι να καταβάλουμε προσπάθειες, να αναλάβουμε, το μερίδιο που μας αναλογεί. Στο τομέα λοιπόν αυτό, μέσω της συνεργασίας που έχουμε στο ΝΑΤΟ, αλλά και στις διμερείς επαφές που έχουμε με τις Ηνωμένε Πολιτείε, έχουμε μια έντονη υποστήριξη από την Αμερική, αρκεί βέβαια να καταφέρουμε και εμείς να φτάσουμε σε μια ποιοτική βελτίωση στη δική μας την πλευρά. Μπορώ να επισέλθω σε περισσότερες λεπτομέρειες εφόσον έχετε ερωτήσεις. Προσπαθήσαμε ουσιαστικά να καλύψουμε τις διάφορες πτυχές του ενέργειου ανεφοδιασμού καυσίμων, δηλαδή την διαθεσιμότητα του εξοπλισμού, να γίνει δηλαδή η απαραίτητη αγορά εξοπλισμού. Υπάρχει εξοπλισμός που αγοράζεται από τα κράτη-μέλη το 400 μη το MRTT της Airbus, επίσης είναι το Multi Role Tanker Transport, είναι ένας άλλος εξοπλισμός ο οποίος μπορεί να αγοραστεί από τα κράτη-μέλη, είτε μπορεί να δοθεί στα κράτη-μέλη με τη μορφή παροχής υπηρεσίας από το ένα κράτος μέλος στο άλλο. Δηλαδή ένα κράτος μέλος θα μπορούσε, ορισμένα κράτη-μέλη είπανε ότι μπορούν να αγοράσουν έναν εξοπλισμό, άλλα κράτη-μέλη είπαν ότι μπορούν να παρέχουν συγκεκριμένε υπηρεσίε. Το ίδιο και για το 400 μη. Ορισμένα κράτη-μέλη θα έχουν το σκάφος αυτό, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον αέριο εφοδιασμό. Θα μπορούσαμε στη συνέχεια, εφόσον εντοπίσουμε τα κράτη-μέλη που θα έχουν το σκάφος αυτό, να δημιουργήσουμε ένα συμπληρωματικό δίκτυο εφοδιασμού, να καλύπτει και τα κράτη-μέλη αυτά που δεν θα έχουν αγοράσει το αεροσκάφο. Πρέπει όμως να μας απασχολήσει και το ζήτημα της απασχόλησης μετά, προκειμένου να έχουμε και κοινά προγράμματα συντήρησης, κατάρτισης, προκειμένου να καταφέρουμε αποτελεσματικά όλοι να χρησιμοποιήσουμε τα αεροσκάφη αυτά. Και ουσιαστικά εδώ πέρα βασιζόμαστε στη γνώση που υπάρχει ήδη στα πλαίσια του ACT όσον αφορά την ε, κοινή διοικητική μέρημνα για τα αεροσκάφη. Τέσσερα κράτη-μέλη αυτή τη στιγμή έχουν αρχίσει να συμμετέχουν και τα κράτη αυτά μέλη ήδη έχουν αρχίσει να βοηθούν άλλα κράτη-μέλη, παρέχοντά τους συγκεκριμένες υπηρεσίες. Δεν περιμένουμε όμως τη στιγμή αυτή που θα παραδοθούν τα 400M και τα MRTT. Ήδη κάνουμε κάποια πράγματα. Για παράδειγμα, η Ιταλία ήδη έχει τη δυνατότητα ανεφοδιασμού μέσω αεροσκαφών Boeing. Επομένως, έχει ήδη αρχίσει η Ιταλία να βοηθά και άλλα κράτη-μέλη να χρησιμοποιούν τις δικές ουσιαστικά τις στρατιωτικές δυνατότητες. Προσπαθούμε δηλαδή ήδη με αυτά που έχουμε να καλύψουμε τις ανάγκες μας μέσω πρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Σας ανέπτυξα τώρα ένα παράδειγμα λίγο περισσότερο. Το ίδιο θα μπορούσα να κάνω και με άλλα παραδείγματα. Όπως για παράδειγμα τις ασκήσεις που γίνονται όσον αφορά την κατάρτιση πιλωτών ελικοπτέρου θεωρώ ότι είναι ένα από τα καλύτερα παραδείγματα που έχουμε στα πλαίσια της συνεργασίας στο ΝΑΤΟ. Τα κράτη-μέλη εποφελούνται τέτοιων προγραμμάτων κατάρτισης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στη συνέχεια ακόμα και σε αποστολές του ΝΑΤΟ, όπως για παράδειγμα στο Αφγανιστάν, είναι σε θέση να παρέμβουν χρησιμοποιώντας την εμπειρογνωμοσύνη αυτή που έχουν κερδίσει. Την προηγούμενη εβδομάδα το Βέλγιο, στο Κλάνιμπεργκεν, δεν ξέρω αν το πρόφερα σωστά, υπήρχε ένα κοινό πρόγραμμα κατάρτισης για πληρώματα ελικοπτέρου που συμμετείχαν άνθρωποι από το Βέλγιο, την Ιταλία, τη Γερμανία και την Ισπανία μαζί με τις ειδικές βελγικές δυνάμεις, τόσο τις στρατιωτικές όσο και τις αστυνομικές. Το ίδιο έχει γίνει και για, τους, και για τα πυρομαχικά, το ίδιο έχει γίνει και για τις α, κινητές αυτές κλινικές στην Ήπεθρο, τις οποίες ανέφερα. Το ίδιο έχει γίνει και στα πλαίσια του pooling and sharing. Όσον αφορά ένα πρόγραμμα της που υπεγράφει την προηγούμενη εβδομάδα από πέντε κράτη-μέλη, προκειμένου να μπορούν τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να έχουν κοινή πρόσβαση σε ένα δορυφορικό πρόγραμμα σε χαμηλότερες τιμές, προκειμένου να καταφέρουν να αποκριθούν στις επιχειρησικές τους ανάγκες. Δεύτερον, αναφερθήκατε στον κώδικα συμπεριφοράς. Ξέρετε ότι στα πλαίσια του pooling and sharing αναφερόμαστε γενικότερα στην συνένωση και κοινή χρήση του στρατιωτικού δυναμικού που θα λειτουργήσει όμως εφόσον τα κράτη-μέλη εθελοντικά εντελώς αποφασίσουν να συμμετέχουν. Δεν θα περάσω αυτή τη στιγμή σε πάρα πολλέ λεπτομέρειε. Θέλουμε βασικά να έχουμε 10 περίπου αρχές σε σχέση με τις οποίες θα δεσμευτούν εντελώ εθελοντικά τα κράτη-μέλη, προκειμένου να υπάρχει μια μακροπρόθεσμη και διαρθρωμένη συνεργασία στα πλαίσια του pooling and sharing. Ορισμένα κράτη-μέλη το έχουν κάνει ήδη, όπως η Σουηδία. Αυτό που θέλουμε είναι να χρησιμοποιηθούν περισσότερο οι πρακτικές αυτές και κάτι ακόμα το οποίο θέλω να αναφέρω είναι ότι πρέπει να γνωρίσουμε ότι το pooling and sharing θα εφαρμοστεί κυρίως σε διμερή περιφερειακή βάση μεταξύ δύο-τριών κρατών μελών, ενδεχομένως και περισσότερα, ενδεχομένως να φτάσουμε τα πέντε και τα έξι κράτη. Πάντως, σε ένα αρχικό στάδιο, ορισμένα μόνο κράτη-μέλη θα συμμετέχουν για τα πιο σημαντικά προγράμματα. Στα πλαίσια της συνεργασίας που έχουμε στην ACT, αυτό ακριβώς έχουμε δει και από την πλευρά του ΝΑΤΟ. Πρέπει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Άμυνας να είναι σε θέση να υποστηρίξει αυτή την διμερή και περιφερειακή συνεργασία και παράλληλα να εξασφαλίσει ότι μπορούμε να έχουμε ένα pooling and sharing à la carte, αυτό είπαν άλλωστε και οι υπουργοί στη Λευκοσία, αλλά παράλληλα να υπάρχει και μια γενικότερη συνεκτικότητα, δηλαδή μια ευρύτερη ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών ανάμεσα σε αυτές τις διαφορετικές ομάδες συνεργασίας, προκειμένου να αποφύγουμε επικαλύψεις, προκειμένου να μην χάνονται κάποιες βέλτιστες πρακτικές προκειμένου να καταφέρνουμε να καλύπτουμε όλες, όλα τα κενά τα οποία ενδεχομένως υπάρχουν χωρίς να έχουμε ιδιαίτερη προστιθέμενη αξία σε έναν μόνο τομέα. Βασίζομαι λοιπόν πάρα πολύ σε αυτή τη διμερή περιφερειακή συνεργασία προκειμένου να στεφθεί με επιτυχία το pooling and sharing. Και Όλοι οι υπουργοί οι οποίοι συμμετείχαν ε, στην ε, άτυπη σύνοδο όντως υποστήριξαν την προσέγγιση αυτή και έπειτα σε επίπεδο ομάδας εργασίας με τους ε, συνήθεις συμμετέχοντες στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Άμυνες και αυτοί με τη σειρά τους εξέφρασαν την ίδια υποστήριξη. Πιστεύω λοιπόν ότι μπορούμε μέχρι την επόμενη συνεδρίαση των Υπουργών που θα λάβει η χώρα το... στις 26 Νοεμβρίου να έχουμε καταλήξει ένα συγκεκριμένο θετικό αποτέλεσμα. Τώρα, για ποιο λόγο η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Άμυνα αποτελεί τελικά την τέλεια πλατφόρμα προκειμένου να ελοποιηθεί το pooling and sharing. Το εξηγείτε εσεί, Πρόεδρε, πάρα πολύ καλά στη δική σα την έκθεση. Εγώ θα επιμείνω σε τρία μόνο σημεία. Καταρχά, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Άμυνα ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επομένω, υπάρχουν όλα αυτά τα στοιχεία συνεργασία προκειμένου να υλοποιηθεί το pooling and sharing. Δεύτερον, έχουμε το δεύτερο αυτό πλεονέκτημα της συνεργασίας που θα τη συνεργασία με τον κοινό οργανισμό συνεργασία στον τομέα των εξοπλισμών. Είναι πάρα πολύ σημαντική η συμφωνία αυτή που έχουμε υπογράψει ακόμα και στην, στον αναέριο εφοδιασμό. Μπορούμε να συνεργαστούμε με την ε, ΟΚΑΡΑ για 400M για το, R, για το MRTT επίσης. Ενδεχομένως ο κύριος Χούιμπρετς να αναφερθεί στα σημεία αυτά πολύ περισσότερο. Το ίδιο ισχύει για την BioDep, για το πρόγραμμα βελτίωσης και ενίσχυσης του βιολογικού εξοπλισμού. Το ίδιο ισχύει και για τα μέτρα τα οποία πρέπει να ληφθούν για τις θαλάσσιες νάρκες. Το σημαντικό είναι να καταλάβουν όλα τα κράτη-μέλη ότι δεν είναι μια τυπική απλώς συμφωνία, είναι μια συμφωνία που πραγματικά θα τροποποιήσει τον τρόπο εργασίας μας. Η συμφωνία αυτή επίσης θα βελτιώσει πάρα πολύ την τεχνολογία και τη βιομηχανία στον τομέα της άμυνας. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Άμυνας βρίσκεται σε συνεχή επαφή με τους συναδέλφους από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θέλουμε να υπάρχει και στον τομέα της βιομηχανίας της άμυνας ένας συντονισμό μεταξύ των κρατών μελών τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόεδρο, σα ευχαριστούμε. Κύριε Χουιμπρέκτς, είστε αναπληρωτή Διευθυντή ε, του Κοινού Οργανισμού συνεργασία στον τομέα των εξοπλισμών. Η ε, ΟΚΑΡΑ ασχολείται με το πρόγραμμα Α400M, με τι φρεγάτες ΦΡΕΜ, με τα ελικόπτερα ΤΙΓΡ, Tiger καθώς επίσης με κάποιους ε, ακόμα πολύ σημαντικούς αμυντικούς εξοπλισμούς θα μας πείτε εσείς τώρα για ποιο λόγο η συμφωνία που έχετε υπογράψει με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Άμυνας θα αποτελέσει κατά τη δική σας άποψη μια ιδιαίτερα θετική εξέλιξη. Σας ευχαριστούμε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Χαίρομαι ιδιαίτερα που, βρίσκεστε, που βρίσκομαι εδώ σήμερα ανάμεσά σας ε, και με την κυρία Αρνό από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Άμενος και να σας πω λίγα στοιχεία για τη συνεργασία μα και γιατί αυτή η συμφωνία που υπογράψαμε είναι τόσο σημαντική τα βασικά έργα της ΟΚΑΡ είναι να κάνει διαχείριση ε, προγραμμάτων ε, άμυνας ε, σε συνεργασία. Για να μπορέσουμε όμως να διαχειριστούμε αυτά τα προγράμματα, όλα αυτά θα πρέπει να ενταχθούν στον ΟΚΑΡ, διότι ο ΟΚΑΡ είναι ένας ανεξάρτητος διεθνής οργανισμός με τους κανόνες του και η βασική δυσκολία ένταξης προγραμμάτων είναι η εναρμόνιση αρκετών πτυχών, ε, εναρμόνιση απαιτήσεων, χρονοδιαγραμμάτων και προπολογισμών. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι η εναρμόνιση αυτή αποτελεί το επίκεντρο των εργασιών της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Άμενας. Γι' αυτό και μας, μας χαροποιεί το γεγονός ότι έχουμε ως εταίρο μας ε, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Άμυνας, διότι ουσιαστικά είναι ε, ανώτερη από εμά, είναι πάνω από εμά και μπορούμε να συνεργαστούμε ε, απευθείας για τα θέματα αυτά. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα λοιπόν ε, για την ε, συμφωνία ε, που κάναμε με την Ευρωπαϊκή Ένωση για να στηρίξει την εταιρική μας σχέση, η οποία φυσικά επισημοποιεί την εταιρική σχέση την οποία είχαμε ε, στην πράξη εδώ και αρκετό καιρό. Τώρα όμως λαμβάνει και την προβολή που της αξίζει αυτή η εταιρική σχέση. Στόχος μας είναι ακριβώς να εφαρμόσουμε αυτή τη συνεργασία πλήρως ε, και να υπάρχουν διαπαφές ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Άμυνας και ο ΚΑΡ, να λειτουργούν αυτές όσο πιο αποτελεσματικά γίνεται και να έχουμε και αποτελέσματα. Και τα αποτελέσματα φυσικά είναι αυτά τα συγκεκριμένα προγράμματα ε, στα οποία αναφέρθηκε ήδη η κυρία Αρνό, εντός ε, των πρωτοβουλειών pooling and sharing και φυσικά Υπάρχουν και κάποια εξαιρετικά παραδείγματα. Υπάρχει ένα πρόγραμμα το οποίο αποκαλείται MOPCM, ε, τα οποία είναι ε, θαλάσσια μέτρα, ε, τα οποία αναπτύσσονται αυτή τη στιγμή και ενσωματώνονται στο ΝΟΚΑΡ για θαλάσσιες νάρκες και έτσι συνεργαζόμαστε, εντάσσουμε τα στοιχεία αυτά και πάντα το έργο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Άμυνας είναι πολύ ευρύτερο από το δικό μας. Εμείς ε, είμαστε περιορισμένοι σε συγκεκριμένα ε, κράτη-μέλη που συμμετέχουν ε, σε συγκεκριμένα προγράμματα. Υπάρχει επίσης και το Musis, που έχει συγκεκριμένα συστήματα παρατήρησης, χερσαία, και υπάρχει και το ESOR, το οποίο είναι το European Secured Software Radio, ένα πρόγραμμα το οποίο έχει πολύ περιορισμένο πεδίο εφαρμογή. Έχουμε έξι κράτη που συμμετέχουν σε μία φάση του προγράμματος και έχουμε και το Music το οποίο στο μέλλον συμμετέχει σε ευρύτερο πρέσιο και προσπαθούμε να δούμε ποιο είναι το πραγματικό πεδίο εφαρμογή του προγράμματο Μπορούμε να σας απαντήσουμε σε όλες μας τις ερωτήσεις όταν θα επισέλθουμε στις λεπτομέρειες. Ευχαριστώ. Υπάρχουν συνάδελφοι που θέλουν να πάρουν τώρα το λόγο, συνάδελφοι που επιθυμούν διευκρινήσεις. Άντριο. Yes, uh, good afternoon. I... Ε, καλησπέρα σας. Ζητώ συγγνώμη γιατί χρειάστηκε να βγω λίγα και μάλλον μου διέφυγε κάτι. Αλλά έχω την εντύπωση πως πολύ τεχνική ε, συνεργασία. Καλή είναι και βελτιώνεται. μεταξύ ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκής Ένωσης και η υπηρεσία παίζει μεγάλο ρόλο. Η πολιτική συνεργασία ε, είναι μεταβίας αντιληπτή και αναρωτιέμαι εάν η κυρία Αρνό βρίσκει την έλλειψη πολιτικής ε, διάστασης στην προσπάθεια βελτίωσης ε, της ε, ενοποίησης του στρατιωτικού συμπλέγματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης αν θεωρεί πρόβλημα. Το δεύτερο ερώτημα αφορά τη συγχώνευση των δύο εταιριών της EADS και της British Aerospace. Δεν θεωρείτε πως αυτό σε μία μέρα θα έκανε πολύ περισσότερα όσον αφορά την ενοποίηση των ενόπλων δυνάμεων και των δυνατοτήτων τους από χρόνια ολόκληρα δουλειάς ε, της ε, υπηρεσίας άμυνας και θεωρείται την υπηρεσία άμυνας πως η δουλειά σας αξιολογείται και εκτιμάται από τα κράτη-μέλη. Θα μπορούσαν να εκμεταλλευθούν την έξοχη εργασία σας καλύτερα από όσο το κάνουν. Εάν υπήρχε η πολιτική βούληση να εμπιστευθούν αλλήλους και η έλλειψη εμπιστοσύνης μπορεί να αντιμετωπιστεί από τις αλλαγές στον τομέα των, των επιχειρήσεων των αμυντικών. Ευχαριστούμε. Απαντώντας σε κάποιες από τις ερωτήσεις του Άντριου, χωρίς όμως να θέλω να φέρω σε θέση τους προσκεκλισμένους μας, διαβάσαμε ότι ορισμένοι Υπουργοί Άμυνας μιλήσανε με πολύ ανοιχτό πνεύμα στον τύπο και δεν ήταν πάρα πολύ ενθουσιώδης τελικά για το pooling and sharing ήταν απλώς ε, εκνευρισμένοι, ενδεχομένως να μην κατάλαβαν καλά πώς θα λειτουργήσει το, πρόβλημα, το πρόγραμμα, με συγχωρείτε, ή τελικά καταδεικνύουν οι δηλώσεις αυτές ότι υπάρχει τελικά ένα μεγάλο χάσμα ανάμεσα στα κράτη-μέλη και ότι τελικά δεν έχει γίνει απόλυτα κατανοητή διαφορά ανάμεσα στο pooling and sharing και το smart defense. Merci. Uh, Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τον κύριο Ντάφ. Και για τις ερωτήσεις του. Για τη συνεργασία τώρα με τον ΝΑΤΟ. Ναι, υπάρχει πολύ καλή συνεργασία στο τεχνικό επίπεδο. Δεν μπορώ να πω πως όλα έχουν λυθεί στο θεσμικό επίπεδο. Έχουμε πολύ ακόμα και βέβαια καλύτερο θα ήταν να δούλευαν τα πράγματα και στο τεχνικό επίπεδο και να έχουμε και μια άλλη θεσμική τάξη που δυσκολεύει το πολιτικό επίπεδο. Βεβαίως, καλό θα είναι μια μέρα να υπάρξει μια λύση στο πολιτικό επίπεδο και ό,τι συνεισφέρει σε αυτό βεβαίως είναι δεκτό. Το γεγονός πως εργαζόμαστε καλά στο τεχνικό επίπεδο και ότι βεβαίως είμαστε ανοιχτοί και σε συμμάχους εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι σημαντικό. Η ποιότητα νομίζω της ε, συνεργασίας είναι κάτι το οποίο καθιστά τις ευρωπαϊκές προσπαθίες πιο σημαντικές ε, και για τη ΣΥΠΑ. Και νομίζω θα υπάρξει και συστηματική συνεργασία ε, με τον Καναδά και για τους μη Ευρωπαίους, ειδικά τους πέραν του Ατλαντικού. Έχει νόημα αυτή η τεχνική συνεργασία και διαβάστε τη δήλωση του Σικάγου σε επίπεδο Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ καλωσορίζουν τη συνεργασία και στον τομέα της, ε, του εναέριου ανεφοδιασμού. Και μπορεί να υπάρξει νομίζω και κάποια πολιτική διάσταση από το πώς ε, καλωσορίζεται η τεχνική συνεργασία στην άλλη όχθη του Ατλαντικού. Όπως φαντάζεστε δεν θα σχολιάσω τη συγχώνευση των δύο εταιριών. Αυτό είναι απόφαση των αρμοδίων αρχών. Δεν είναι η δικιά μας δουλειά. Εμείς πάντα λέγαμε πως πρέπει να υπάρχει λιγότερος κατακαιρματισμός, αλλά είναι επίσης σαφές πως το βιομηχανικό τοπίο είναι κατακαιρματισμένο. Πέρα από αυτό δεν έχω τίποτα να πω. Και πάλι αυτό είναι δουλειά των αρμοδίων αρχών. Τώρα το αν το αξιολογούν σωστά τα κράτη-μέλη, τη δουλειά μας δηλαδή, και αν την εκμεταλλεύονται καλύτερα, θα μπορούσαν. Δεν ναι, θα έλεγα. Και ίσως. Αυτό να οφείλεται στη θετική ατμόσφαιρα. Πως ε, ήταν ε, δύο υπουργοί στην, ε, στην Κύπρο. Η άμυνας που έκανε πολύ καλές συζητήσεις, τα εξήγησε ο Ματσικοπόφσκι και στον τομέα των δυνατοτήτων και όσο περισσότερο οι υπουργοί θα συζητάνε ε, πραγματικά τέτοια πράγματα τόσο καλύτερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουμε ευθύνη ως Ευρωπαϊκή Υπηρεσία να φέρνουμε αυτά τα πράγματα στο υπουργικό επίπεδο και να τους βάζουμε σε μια θέση ώστε να μπορούν να δώσουν πολιτική όθηση στις ομάδες τους. Και νομίζω πως το δυσκολότερο δεν είναι η πολιτική βούληση στο επίπεδο των Υπουργών, αλλά αφορά παλαιούς κρατεούς μηχανισμούς ε, στα κράτη-μέλη, γραφειοκρατίες, ε, που, που πρέπει να αντιληφθούν πως η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία μας έχει προσθέμενη αξία, γιατί ειδικά στα μεγαλύτερα κράτη-μέλη. Έχουμε μηχανισμούς που λειτουργούν καλά και αντιμετωπίζουν αυτή τη στιγμή δυσκολίε με την οικονομική κρίση. Η πρώτη του αντίδραση δεν είναι να πούν πω θα λύσει τα προβλήματά μας αυτή η υπηρεσία, όχι ότι θα τα λύσουμε. Αλλά παρόλα αυτά, νομίζω πως υπάρχει μια προσθέμενη αξία. Και ναι, νομίζω πως μπορούμε να μπορούν να μας χρησιμοποιήσουν καλύτερα, πρέπει να προσαρμοστούμε και εμείς. Και βέβαια υπάρχουν και κάποια καθήκοντα της υπηρεσίας μας, π.χ. το σχέδιο ανάπτυξης δυνατοτήτων πρέπει να γίνει πιο φιλικό προς τους χρήστες για να ξέρουν καλύτερα το τι συμφωνούν τώρα. Για την έλλειψη εμπιστοσύνη έχετε δίκιο. Όταν κάνει κάποια πράγματα η βιομηχανία σε λίγες ώρες ή εβδομάδες, καλά καμιά φορά βεβαίω για να εφαρμοστούν αυτά τα πράγματα χρειάζονται χρόνια, αλλά δημιουργούν αυτή την εμπιστοσύνη και αυτό είναι σημαντικό στοιχείο. Επίσης αυτό το οποίο κάνουμε στον τομέα της εκπαίδευσης είναι πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο εμπιστοσύνης. Πρέπει να πω πως Η αξιωματική όταν συμμετέχουν σε ασκήσεις όπως αυτή που έγινε πριν από μια εβδομάδα ε, στην Πορτοκαλία, στο Βέλγιο, ε, είναι ζήτημα εμπιστοσύνη. Οι στρατιωτικοί δεν το λένε και φιλία ακόμα. Είναι δηλαδή οι άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται στο πεδίο και αναπτύσσουν μια εμπιστοσύνη που βεβαίω είναι απαραίτητη στις ασκήσεις. Οι εκπαιδευτικές αυτές δραστηριότητες λοιπόν Ακόμα και το ότι μπορούμε να έχουμε κάποια αμοιβαία αναγνώριση των διαδικασιών της εκπαίδευσης, ε, μια κοινή διδακτέα ύλη, να είναι νομίζω μια αρχή, θα έλεγα, της εμπιστοσύνης, ε, το οποίο δεν υποβάζω καθόλου. Η ερώτηση του Προέδρου για κάποια επιφυλακτικότητα, η ενόχληση από κάποιους υπουργούς για την κοινή χρήση του υλικού. Για τους υπουργούς που λένε πως όλα αυτά τα πράγματα λέμε, pulling and sharing, smart defense, νομίζω πως η, μια πρώτη επιφύλαξη που υπάρχει. Ε, Συνεχίζω στα γαλλικά. Μία επιφύλαξη λοιπόν όσον αφορά το pooling and sharing, γιατί ζητήσαμε από τα κράτη-μέλη παράλληλα να συμμετέχουν στο pooling and sharing και από την άλλη να μειώσουν τους προπολογισμούς τους. Αν ουσιαστικά το pooling and sharing αποτελεί άλοθη για να μειωθούν οι αμυντικοί προπολογισμοί, τότε καταλαβαίνω τις επιφυλάξεις των Υπουργών. Το pooling and sharing δεν σημαίνει ότι θα κάνουμε περισσότερα πράγματα έχοντας λιγότερα. Θέλουμε να πετύχουμε περισσότερα πράγματα με αυτά τα οποία πρέπει να διαθέτουμε. Υπάρχουν ορισμένοι υπουργοί που φοβούνται ότι θα χρησιμοποιηθεί το pooling and sharing ως άλοθη για να μειωθούν οι αμυντικοί προπολογισμοί και ότι στο όνομα τελικά της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας θα μειώσουμε τελικά τους εξοπλισμούς στο στρατικό δυναμικό ενώ ουσιαστικά το αντίθετο ακριβώς απαιτεί διεθνής κατάσταση. Πρώτον αυτόν. Δεύτερον, μας λένε μερικές φορές ότι έρχεστε εσείς, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Άμυνας, με όλα αυτά τα κράτη-μέλη τα οποία εκπροσωπείτε και μέσω της ομοφωνίας σας τελικά καθιστάτε τα πράγματα ακόμα πιο πολύπλοκα. Αυτό που θέλουμε να δείξουμε δεν αληθεύει κάτι τέτοιο. Με τη συνεργασία δύο κρατών μελών μπορούμε να έχουμε μια πάρα, ένα πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα. Πολλές φορές, βασιζόμενοι απλώς σε μια περιφερειακή συνεργασία, μπορούμε να έχουμε ένα αποτέλεσμα ιδιαίτερα θετικό, το οποίο θα είναι σε θέση να εφαρμόσουν και άλλα κράτη-μέλη στη συνέχεια. Αυτό ακριβώ θέλουμε να προωθήσουμε ω Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Άμυνα, ξεκινώντα από μια διμερή περιφερειακή συνεργασία να δημιουργήσουμε βέλτιστε πρακτικέ. Δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε επιπλέον γραφειοκρατικό ακθο Αυτό που θέλουμε είναι να βοηθήσουμε τα κράτη-μέλη να έχουν πρόσβαση σε συγκεκριμένες μελέτες που έχουν γίνει. Ο κύριος Χάιμπρεκτς αναφέρθηκε επίσης στις θαλάσσιες νάρκες και κυρίως στα μέτρα τα οποία θα πρέπει να ληφθούν κατά των αρκών αυτών. Υπάρχουν κράτη-μέλη όπως οι Γάλλοι και οι Βρετανοί, οι οποίοι αποφάσισαν διμερώς να ασχοληθούν με το ζήτημα αυτό. Επιλήφθηκαν λοιπόν του ζητήματος και πολύ γρήγορα κατάφεραν να καλύψουν τις δικές εθνικές ανάγκες και δώσαν έπειτα την τεχνογνωσία τους αυτή στον ΟΚΑΡ προκειμένου να χρησιμοποιηθεί και από άλλα κράτη-μέλη. Έχετε λοιπόν ήδη μια πάρα πολύ καλή πλατφόρμα, μια ήδη πολύ καλή εμπειρογνωμοσύνη η οποία υφίσταται, η οποία δεν περιπλέκει τα πράγματα, δεν δημιουργεί επιπλέον διαδικασίες, αλλά αντίθετα απλοποιεί τη συνεργασία η οποία πρέπει να υπάρχει ανάμεσα στα κράτη-μέλη και στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Άμυνας. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικές οι εμπειρίες αυτές και δεν θα πρέπει να τις υποτιμούμε. Βάσει τα όσα είπατε στην πρώτη σας απάντηση, οι ε, υπουργοί οι αρμόδιοι του προπολογισμού ανήκουν και αυτοί στους συνομιλητές σας ή περιορίζετε μόνο στους υπουργούς άμυνας. Κοιτάξτε, δεν ανήκουν στην άμεση αρμοδιότητά μου, ούτε συμμετέχουν σε κάποιο συμβούλιο, πάντως τους έχουμε συνεχώς κατά νου. Οι Υπουργοί Άμυνα έχουν πάντα κατά νου αυτά τα οποία του λένε οι Υπουργοί που είναι αρμόδιοι για του προπολογισμού. Και θεωρώ ότι και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Άμυνα μπορεί να αποτελέσει ένα χώρο μέσω του οποίου και οι Υπουργοί που είναι αρμόδιοι για του προπολογισμού μπορούν να εκθέσουν τις δικές τους ιδέες, ιδίω όταν θέλουν να διατηρήσουν κάποιες πιστώσεις ή να μας δείξουν σε ποιους τομείς μέσω της συνεργασίας έχουν καταφέρει να κάνουν εξοικονόμηση. Ο κύριος Αντιπρόεδρος έχει το λόγο, παρακαλώ. Μια ερώτηση προς την κυρία Ναρνού. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία, όπως έχει λεχθεί από εσά, ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση εθαρρύνει την εμπλοκή των κρατών μελών για να συμμετέχουν. Έχει συνεργασία με τις ΗΠΑ και τον Καναδά. Η αμυντική βιομηχανία επίσης συνεισφέρει. Και βέβαια πρέπει να αναζητηθεί ένας καλύτερος τρόπος, τρόπος συντονισμού μεταξύ των κρατών που συμμετέχουν. Δύο συγκεκριμένες ερωτήσεις. Μέσα από τη διαπίστωση ότι υπάρχουν κράτη-μέλη που ανήκουν και στο ΝΑΤΟ αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, νομίζω εκεί είναι σαφές ότι υπάρχει κοινό στόχος και τόπος. Το ερώτημα που θέτω προς εσάς είναι ποια είναι η αντίδραση των κρατών που ουσιαστικά συμμετέχουν μόνο στο ΝΑΤΟ ή μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αν μέσα από τις όποιες αντιδράσεις τους και είναι εσείς θα μας πείτε βοηθούν την προσπάθεια σας διότι εδώ είναι το σημαντικό και το δεύτερο έχετε κάνει μια αναφορά για τις Ηνωμένε Πολιτείε, όπου έχετε μια συνεργασία και με τον Καναδά, ειδικότερα για τις Ηνωμένε Πολιτείε. Και εκτιμώ ότι το πολιτικό ερώτημα που πρέπει να σταθείτε και να απαντήσετε με πιο συγκεκριμένο τρόπο δεν είναι αν έχουμε συνεργασία με τις Ηνωμένε Πολιτείε, αλλά τι απαιτούν οι Ηνωμένε Πολιτείε, γιατί κάνατε μια αναφορά, από τα κράτη-μέλη που συμμετέχουν. Επιβάλλουν άποψη ή απλώς τοποθετούνται, αν μου επιτραπεί έκφραση, χαλαρά. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ζητώ συγγνώμη, έχασα την αρχή της παρέμβασής σας γιατί δεν είχα φορέσει εγκαίρως τα ακουστικά. Πάντω, αν να παραλείψω κάτι στην απάντησή μου, ευχαρίστως να μου πείτε τι παρέλειψα. Τώρα, όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ. Κοιτάξτε, ακριβώς επειδή υπάρχουν διαφορές, γι' αυτό το λόγο είναι πολύ σημαντική και η συνεργασία. Θέλουμε προφανώ μέσω του ΝΑΤΟ να έχουμε μια συμμαχία και μια συνεργασία με τι Ηνωμένε Πολιτείε τον Καναδά, καθώ επίση και με άλλε χώρε οι οποίε βρίσκονται στην Ευρώπη, ενδεχομένω να μην συμμετέχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επομένω, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ καλό το ότι μπορούμε και έχουμε αυτή την διατλαντική σχέση στα πλαίσια του ΝΑΤΟ. Και είναι πολύ θετικό επίση το ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε χώρε που δεν ανήκουν στο ΝΑΤΟ επειδή έτσι επέλεξαν από πολιτικής πλευράς χώρες όμως οι οποίες είναι σημαντικοί παράγοντες όσον αφορά τη διαχείριση των κρίσεων. Αναφέρομαι για παράδειγμα στις σκανδιναβικές χώρες που δεν συμμετέχουν στο ΝΑΤΟ. Αναφέρομαι επίσης στην Αυστρία, στην Ιρλανδία που συμμετέχουν πάρα πολύ στη διαχείριση των κρίσεων. Θεωρώ λοιπόν ότι το όλο σύστημα ως έχει αλλοσυμπληρώνεται πολύ καλά. Υπάρχουν βέβαια ορισμένα κράτη-μέλη τα οποία βρίσκονται στο ΝΑΤΟ και όχι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το αντίστροφο μπορείτε εύκολα να φανταστείτε σε ποιον αναφέρομαι, σε ποια κράτη αναφέρομαι. Ναι, όντως, εκεί πέρα μπορεί να υπάρχει ένα πρόβλημα. Δεν νομίζω όμως ότι αυτό το ειδικό πρόβλημα το οποίο μπορεί, ελπίζω, να επιληθεί πολιτικά στο άμεσο μέλλον, δεν θα πρέπει αυτό το πρόβλημα να μας κάνει να ξεχνάμε ότι είναι πάρα πολύ θετικό το ότι έχουμε μία διατλαντική συμμαχία με τις Ηνωμένε Πολιτείες και με τον Καναδά και κατά αυτόν τον τρόπο αποφελούνται πολλά κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα οποία έχουν αποφασίσει να μην συμμετέχουν στο ΝΑΤΟ και παρόλα αυτά όμως επενδύουν πάρα πολύ στη διαχείριση των κρίσεων. Όσον αφορά τώρα τις Ηνωμένε Πολιτείε. Αναφερθήκατε στις Ηνωμένε Πολιτείε και στον Καναδά. Ξεκινάμε με τις Ηνωμένε Πολιτείε. Τι περιμένουν από εμά, τι απαιτούν από εμά. Κοιτάξτε, νομίζω το έχουν πει ξεκάθαρα. Ο κύριο Γκέιτς το είπε ξεκάθαρα, ο κύριο Πανέτα επίση και επαναλήφθηκε ακριβώς με τον ίδιο τρόπο στην στρατηγική τους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι security provider, όπως είπανε, επομένως θα πρέπει να συμβάλλουμε στην ασφάλεια και να επομισθούμε το μερίδιο το οποίο μας αναλογεί οι συνομιλητές μας από τις ΗΠΑ Πολιτείες χρησιμοποιούν και κάποιες λέξεις που δεν θα περιμέναμε πριν από μερικά χρόνια. Μας λένε να είστε έτοιμοι να επέμβετε αυτόνομα. Be autonomous μας λένε. Μην επαφίεστε μόνο σε εμά για να κάνουμε το 80%. Σε κάποιες περιπτώσεις θα το κάνουμε, σε άλλες πάλι όχι. Και είναι φυσιολογικό αυτό το πράγμα. Γιατί ουσιαστικά το βάρος βρίσκεται αλλού γιατί η πρόκληση για τη διατήρηση της ασφάλειας βρίσκεται αλλού και ουσιαστικά εναπόκειται σε εσά, Ευρωπαϊκή Ένωση, να αναλάβετε μεγαλύτερο μερίδιο. Οι Ηνωμένε Πολιτείε που μα λένε είναι do more, κάντε περισσότερα. Uh, να προσθέσω απλώς ότι εμείς θα μπορούσαμε να δεχτούμε αυτή την ενδεχόμενη κατάσταση συνεργασίας όπου θα υπάρχει συνεργασία εντός του προγράμματος με την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο εάν τα κράτη μας αποφασίσουν ότι η ομάδα των χωρών που συμμετέχει ε, μπορεί να συμπεριλαμβάνει και τη ΣΥΠΑ και τον Καναδά και να υπάρχουν ωφέλη σε αυτή την περίπτωση και τότε θα μπορέσουμε να συνεργαστούμε. Δεν έχω τίποτα άλλο να προσθέσω. Ευχαριστώ. Uh, Άλλοι συνάδελφοι θέλουν να πάρουν το λόγο. Υπάρχουν ερωτήσεις ή παρατηρήσεις. Αν όχι, τότε έχουμε σεβαστεί απόλυτα το χρόνο που είχαμε στη διάθεσή μας. Σας ελευθερώνουμε λοιπόν, όπως μας είπατε, την ώρα που ζητήσατε. μισή ακριβώς. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήταν πολύ χρήσιμο πραγματικά να σας ξαναδούμε για να μας πείτε πώς εξελίσσονται γενικότερα οι πολιτικές αυτές του pooling and sharing, τι πρόοδος έχει σημειωθεί. Ελπίζω να είναι ορατή η πρόοδος αυτή στο άμεσο μέλλον και θα μπορούσατε να αναφερθείτε με μεγαλύτερες λεπτομέρειες σε κάποια συγκεκριμένα προγράμματα. Αναφερθήκατε στην ολόκληρο κατάλογο συγκεκριμένων προγραμμάτων. Θα ήταν πολύ ενδιαφέρον λοιπόν για μας να έχουμε μια κάποια ενημέρωση για το πώς προχωράνε τα προγράμματα αυτά και μία αντιπροσωπεία της Υποπιτροπής μας θα πάει τον Ιανουάριο, δεν κάνω λάθος, στην υπηρεσία σας. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που μας προσκαλέσατε και με ιδιαίτερη χαρά θα μεταβούμε για να σας δούμε. Όσον αφορά αυτά τα οποία είπαμε για τους υπουργού Άμυνας και τους υπουργού Προπολογισμού, είναι πάρα πολύ σημαντικό να γνωρίζετε και να αναγνωρίζετε ακόμα περισσότερο η δράση που επιτελείτε εσείς ως Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Άμυνας. Θα πρέπει δηλαδή Μάλλον, οι εμπειρογνώμονε ήδη στα Υπουργεία Άμυνα γνωρίζουν πολύ καλά τι κάνετε. Δεν συμβαίνει όμω το ίδιο και με άλλου εξωματούχου, όταν βγούμε δηλαδή από τον στενό τομέα τη άμυνα. Και ιδίω όσον αφορά τον τομέα των προπολογισμών, καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και οι ηθήνοντε στον τομέα αυτό να γνωρίζουν τι κάνετε, γιατί οι αποφάσει που λαμβάνετε εσεί επηρεάζουν τελικά του αμυντικού προπολογισμού. Και βέβαια και οι βουλευτέ του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλιο και οι βουλευτέ των Εθνικών Κοινοβουλίων μπορούν πραγματικά να συμβάλλουν στο να προωθήσουν περισσότερο την πολύ θετική εργασία που επιτελείται στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Άμυνα. Μπορούμε και εμεί λοιπόν να επιτελέσουμε, αν μου το επιτρέπετε, τον ταπεινό μα αυτό ρόλο η συνεδρίαση που είχαμε στην Κύπρο με τους συναδέλφους από τα Εθνικά Κοινοβούλια ήταν πάρα πολύ χρήσιμη και νομίζω ότι στα πλαίσια της ε, διακοινοβουλευτικής αυτής επαφής που έχουμε πλέον, δηλαδή σε επαφές που έχουμε τα Εθνικά Κοινοβούλια, πολύ συχνά στις ημερήσιες διατάξεις να μπορούμε να μιλάμε περισσότερο για την δική σας υπηρεσία και να ευαισθητοποιούμε περισσότερο τους εθνικούς μας συναδέλφους για αυτά που εσείς κάνετε στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Άμυνας. Θα ήθελα να κάνω μία παρατήρηση. Συμφωνώ απόλυτα με αυτά τα οποία λέτε όσον αφορά και τα εθνικά κοινοβούλια. Δηλαδή υπάρχουν πολλά εθνικά, μάλλον πολλά εθνικά κοινοβούλια που έχουν επιτροπές άμυνας και τα οποία προσκαλούν εμά εκπροσώπου Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Άμυνα, ή θέλουν να μεταβούν για να μας δούνε στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Άμυνας. Θα ήταν πολύ θετικό να ενθαρρυνθούν οι πρωτοβουλίες αυτές και επίσης να επεκτηθούν και σε άλλους ε, βουλευτές που ασχολούνται για παράδειγμα με, τον, με τα θέματα προπολογισμού και θα ήταν πολύ θετικό να προωθηθεί περισσότερο και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Άμυνα σε επαφές που έχετε εσεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τα Εθνικά Κοινοβούλια. Πρόεδρο, όντω ε, ο Άντριου ασχολείται πάρα πολύ με τη συνεργασία που έχουμε με τα Εθνικά Κοινοβούλια. Δεν είναι πάντα εύκολη η συνεργασία αυτή, πάντως μπορούμε να έχουμε πολύ επικοδομητική συνεργασία και ανταλλαγή απόψεων πραγματικά θα δημιουργήσουν μια προστιθέμενη αξία και να έχουμε και συγκεκριμένες συζητήσεις, να ξεφύγουμε δηλαδή από τις θεωρητικές μόνο τοποθετήσεις. Ελπίζω λοιπόν ότι τους επόμενους μήνες θα έχετε και μία πρόταση επίσκεψης από τα Εθνικά Κοινοβούλια ή ότι θα σας δούμε και εσάς στην επόμενη συνεδρίαση που θα έχουμε στην Ιρλανδία. Σας ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε και τον κύριο Χουι Χουιμπρέχτε και καλή συνέχεια στην εργασία σας. Euh, Μάλιστα. Συνεχίζουμε με την εξέταση των εκθέσεων. Τις εκθέσεις μάλλον του κυρίου Πάσκου για τις ε, ρήτρε για την αμοιβαία άμυνα και την αλληλεγγύη. Το συζητήσαμε και στο παρελθόν εκτενώς το ζήτημα αυτό. Περνάμε στην τελική φάση όπου θα συζητήσουμε τις τροπολογίες. όχι, δεν το προσεγγίζουμε από την ιατρική του πλευρά. Είμαι πολύ πιο αισιόδοξο όταν είπα καταληκτική φάση. Στις 25 Οκτωβρίου θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή και στην Ολομέλεια του Νοεμβρίου θα γίνει τελική ψηφοφορία. Κύριε Πασκού, πώς έχουν τα πράγματα. Η έκθεση ζει και βασιλεύει. Κοιτάξτε, σήμερα έγινε μια ψηφοφορία στην Επιτροπή Συνταγματικών Θεμάτων και θα ακολουθήσει και ψηφοφορία στην Επιτροπή Ελευθεριών και έχουμε έξι τροπολογίες που υποβληθήκαν σκιώδης και νομίζω πως έχουμε 102 τροπολογίες καταφέραμε νομίζω να τις καλύψουμε με έξι συμβιβαστικές η συνεργασία που είχα με τους σκιώδεις συγητές και τους εκπροσώπους ε, των διαφόρων φορέων με τη γενική αυτή αρχιτεκτονική ήταν πάρα πολύ καλή. Ήταν ε, επαγγελματικός ο διάλογος και θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους ε, συμμετείχαν γιατί είναι συλλογική δουλειά. Και εγώ άλλο δεν χρειάζεται να πω. Αν υπάρχουν ερωτήσεις, είμαι σίγουρος ότι ο κύριος Νταφ ε, θα ήθελε να πει και εκείνος κάποια λόγια. Ευχαριστώ πολύ λοιπόν. Ευχαριστώ. Θα δώσω λόγο στον Άντριο Μια που είναι και αυτός στην Επιτροπή Συνταγματικών Θεμάτων και εισηγητή εκεί για την ε, γνωμοδότηση. Ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα ευχαριστήσω τον κύριο Πάσκου γιατί ήταν πραγματικά πολύ συνεργάσιμος, ο, πιο συνεργάσιμος συγητής που έχω δει εδώ και πολύ καιρό και με την καλή την έννοια το λέω αυτό, ως κοπλιμέντο. Και ο κύριος Πάσκου λέει άμα είναι έτσι να, να, να αλλάξω στάση. Νομίζω λοιπόν πως οι έξι συμβιβαστικές ε, προτάσεις του είναι καλές και πετυχαίνουν μια ισορροπία μεταξύ των διαφόρων πολιτικών ομάδων και των ε, συνταγματικών ανησυχιών της Επιτροπής μας για να παίξουμε σωστά τα χαρτιά μας ως Ευρωπαϊκή Ένωση και Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Υπάρχει, θεωρώ, κίνδυνος προσπαθώντας να μην εκθέσουμε τις ε, προφανείς ε, αδυναμίες ε, στις πολιτικές μας, τις διαρθρωτικές και τις αμυντικές. Να πάμε στο άλλο άκρο. Και να αρχίσουμε να λέμε πως έχουμε δυνατότητες οποίες δεν έχουμε. Ελπίζω να τις έχουμε κάποια στιγμή, αλλά αυτή τη στιγμή δεν τις έχουμε. Και είναι δύσκολη η ισορροπία. Ειδικά, ειδικά για το κοινό. Δηλαδή η συζήτηση με την κυρία Αρνού είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα γιατί σαφώς το προφίλ της ευρωπαϊκής αυτής υπηρεσίας ακόμα δεν είναι πλήρες εάν πάνε στην Πάφο και έχουν μια επιτυχή συνάντηση Υπουργέ Άμυνας, αυτό είναι καλό, αλλά για να μεταδοθεί η ιδέα, η εμπειρία ότι υπάρχει μια λέσχη, έχουμε ακόμα δρόμο. Οπωσδήποτε στα εθνικά κοινοβούλια και στον τύπο μας. Έχω τώρα δυσκολία με το σχέδιο έκθεσης όπως προέκυψε από την Επιτροπή Συνταγματικών Θεμάτων και η κυρία Γιαννάκου και εγώ διαφωνούμε αν δε το άρθρο 42.7 το ονομάσουμε ρήτρα αμοιβαία συνδρομής ή αμοιβαία άμυνα, εγώ είμαι υπέρ του πρώτου. Γιατί είναι κάτι που αντικατοπτρίζει καλύτερα την συνθήκη, η οποία δεν μιλάει για κοινή άμυνα αλλά ξεκαθαρίζει πως η κοινή ε, άμυνα η χρησιμοποιεί δύο όρους κοινή και συλλογική άμυνα για τη συντριπτική πλειοψηφία της Ένωσης είναι εντός του ΝΑΤΟ και ακόμα και οι χώρες που δεν είναι στο ΝΑΤΟ συνεργάζονται ικανοποιητικά σε τεχνικό επίπεδο εντός του ΝΑΤΟ. και επίσης ως Βρετανός φεντεραλιστής είμαι ιδιαίτερα ευαίσθητος στο φάσμα ενός ευρωπαϊκού στρατού που κυκλοφορεί ειδικά στο εθικιστικό λαϊκιστικό τύπο και δεν θα ήθελα να κάνω κάτι για να έτσι, επιδεινώσω την κατάσταση αυτή. Μια καλύτερη περιγραφή του άρθρου 42.7 είναι μια ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής. Αλλά ε, νομίζω πως τα πράγματα έχουν σήμερα. Τώρα όσον αφορά την ρήτρα αλληλεγγύης, ε, ο κύριος Πάσκου ήταν πάρα πολύ έξυπνος. Μας εξήγησε τι ακριβώ σημαίνει και το τι δεν μπορεί να σημαίνει και βεβαίω τα μελλοντικά βήματα της ε, Κομισιόν και του Συμβουλίου για να οικοδομηθεί ε, αναφέρονται και περιγράφονται πάρα πολύ καλά. Όπως και η διαδικασία λήψης αποφάσεων που πρέπει να ισχύσει στο Συμβούλιο, δηλαδή ειδική ε, πλειοψηφία για τις μη στρατιωτικές πτυχές. Αυτό είναι σημαντικό για εμάς το Κοινοβούλιο, να το τονίσουμε όταν μιλάμε στην Κομισιόν και στο Συμβούλιο όταν θα γίνει αυτό στην Ολομέλεια. Η κυρία Γιαννάκου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, πράγματι όπως ε, σας ανέφερε ο κύριος Πασκού το πρωί ψηφίσαμε την έκθεση DAF δηλαδή ως γνωμοδότηση για, το, ε, για την έκθεση Πασκού και εντάξει υπήρξαν διαφωνίες και είναι φυσικό στη δημοκρατία υπάρχουν διαφωνίες. Αλλά έγινε ψηφοφορία και η άποψη του κυρίου Νταφ δεν έγινε δεκτή. Ο κύριος Πασκού έχει προετοιμάσει μια σειρά τροπολογιών ε, συμβιβαστικών που εμάς μας βρίσκουν σύμφωνους. Τώρα ως προς ε, ορισμένες τροπολογίες ε, του κυρίου Νταφ που δεν μπορούν να περιληφθούν λόγω του διαφορετικού τους περιεχομένου το οποίο είναι ασυμβίβαστο με αυτό που περιλαμβάνουν τροπολογίες είπαμε στη συνάντηση που κάναμε ότι θα πρέπει να ψηφιστούν χωριστά την Επιτροπή μας και όπως αποφασίσει η Επιτροπή επομένως δεν είναι αντικείμενο αν εγώ διαφωνώ με τον κύριο Νταφ. Το αντικείμενο είναι τι αποφασίζει η Επιτροπή, τα δημοκρατικά όργανα. Και αυτό που θα αποφασίσουν, αυτό θα ακολουθήσουμε. Η ουσία είναι όμως ότι η Ευρωπαϊκή Ανώση με τη συνθήκη της Λισαβόνας έχει δική της νομική προσωπικότητα. Και επομένως έχει όλο το δικαίωμα και θα σας έλεγα την υποχρέωση ακόμα κι αν αυτό δεν περιλαμβανόταν στη συνθήκη, να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις προστασίας των πολιτών, όπως σωστά αναφέρεται στην έκθεση του κυρίου Πασκού, και των μελών της. Εάν θεωρήσουμε ότι για να ρυθμιστεί οποιοδήποτε θέμα απειλής, τρομοκρατικής λοιπά η επίθεση από τρίτων εναντίον μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να ερωτήσουμε το ΝΑΤΟ, τότε τι θα κάνουμε για τις χώρες που δεν είναι μέλη του ΝΑΤΟ. Εδώ μιλάμε για μια τελείως διαφορετική αντίληψη και δομή. Άλλωστε προηγουμένως είχαμε συζήτηση για τη συνεργασία επιστρατιωτικών θεμάτων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει προχωρήσει. Τώρα, τα μέλη της Ένωσης που είναι μέλη του ΝΑΤΟ γνωρίζουν τις υποχρεώσεις τους προς τη Συμμαχία και δεν την αμφισβητούν. Ουδής αμφισβητεί την ε, σημασία του ΝΑΤΟ και την παρουσία του εκεί. Δηλαδή ε, καλλιεργείται ο φόβος ότι αν η Ευρώπη προχωρήσει ένα βήμα πιο πέρα θα συμβεί κάτι στο ΝΑΤΟ. Αυτά δεν ισχύουν κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι όλοι μας το γνωρίζουμε, άλλωστε σας θυμίζω ότι στην προετοιμασία που έγινε στην Ευρωπαϊκή Συνέλευση υπήρχε ειδική ομάδα εργασίας υπό τον Επίτροπο Μπαρνιέ η οποία επεξεργάστηκε τα θέματα αυτά. Αποτελούσε δηλαδή αντικείμενο πολιτικό η υπόθεση αυτή. Εάν δεχόμαστε την άποψη του κυρίου Ντάφ, όπως έχει εκφραστεί ιδιαίτερα σε μια τροπολογία, τότε είναι σαν να καταργούμε την έκθεση του κυρίου Πασκού. Κάτι που εμείς δεν το θέλουμε ως Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα εμείς υποστηρίζουμε αυτές τις ενέργειες της Ένωσης, διότι σε τίποτα δεν διακυβεύουν την υπάρχουσα συμμαχία και τις δυνατότητές της και βεβαίως υποστηρίζουμε και την έκθεση του κυρίου συναδέλφου, του κυρίου Πασκού και τις α, συμβιβαστικές τροπολογίες και συμφωνούμε να ψηφιστεί στις 25 του μηνός ε, στο Στρασβούργο. Αυτό είναι ένα πρώτο βήμα κύριε Πρόεδρε που είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί πρόκειται για πολιτική κατεύθυνση και απόφαση και είναι από τα στοιχεία που βασίζονται σε άρθρα της συνθήκης που έχουν πραγματικά αμυγός πολιτικό χαρακτήρα. Δηλαδή τι μπορεί και πρέπει να κάνει ένας διεθνής οργανισμός με το χαρακτήρα που έχει ένωση με πλήθος υπερεθνικών οργάνων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων για την προστασία των μελών της, της κυριαρχίας τους και κυρίως των πολιτών της. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Merci. Σας ευχαριστούμε. Η κυρία Λέζινγκ, σκιώδη συγγήτρια. Ευχαριστώ. Σε μία από τις τελευταίες συνεδριάσεις ανέπτυξα τις επιφυλάξεις μας επί της αρχής για τη φιλοσοφία αυτή αλληλεγγύης και στις δύο περιπτώσεις και στην περίπτωση συνδρομής και στην περίπτωση αλληλεγγύης δηλαδή τη χρήση στο, εσωτερικό. Δεν θέλω να τα επαναλάβω τώρα. Η συζήτηση και η σημερινή συζήτηση έδειξαν πως ε, ακόμα και αν υπάρξουν κάποιες ε, τροπολογίες ε, δεν εκφράζεται η θέση μας. Οπότε θα υποβάλουμε μια έκθεση της μειοψηφίας. Θα ήθελα εγώ να αναφερθώ στην τοποθέτηση της Επιτροπής ΛΥΜΕ όπου αναφέρεται πως ε, εμείς ε, λέμε πως δεν αναφέρεται εδώ πέρα και δεν καθορίζεται παρκώς το πεδίο χρήσης ε, και εφαρμογής αυτής της ρήτρα αλληλεγγύης και νομίζουμε πως στο πλαίσιο της δημοκρατίας θα ήταν καλό να γίνει κάτι τέτοιο. Ευχαριστώ. Ο κύριος Δαφ, ναι. Για τόσα είπε η κυρία Λέζινγκ. Νομίζω ότι είναι πολύ ακριβής ο ορισμός ε, μάλλον ένας πολύ ακριβή ορισμός ε, των συνθήκων ε, βάσει των οποίων θα μπορούσαν να συμβούν ε, κάποια πράγματα δεν είναι σωστός. Βρισκόμαστε σε μία περίοδο που το να το διαμορφώνει τους κινδύνους που αντιμετωπίζουμε, αλλάζει συνεχώς και θα ήθελα να έχουμε μια πιο ελαστική προσέγγιση μια προπτική που θα μας επιτρέπει να είμαστε λίγο πιο ρεαλιστές ε, όταν πρέπει να είμαστε. Η κυρία Γιαννάκου προσδίδει ιδιαίτερη σημασία ε, στο σκεπτικό ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, διαθέτει νομική οντότητα πλέον. Το να διαθέτει κάποιος νομικό πρόσωπο σημαίνει ότι υποχρεούται να σέβεται το γράμμα του διεθνούς δικαίου και να αναγνωρίζει τις δεσμεύσεις των μελών της Διεθνούς Συνθήκης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ναι, είναι πολιτεία. Ελπίζω ότι θα διαμορφωθεί σε πολιτεία. και σε μια πολιτεία που δεν έχουμε τις γενικές αμμοδιότητες και δεν έχουμε κυβέρνηση και δεν είναι αμυντικός οργανισμός. Υπάρχουν άλλες παρεμβάσεις. Ιωάννα. Ευχαριστώ πολύ και πάλι. Σας ευχαριστώ για τη συζήτηση. Δύο σχόλια. Καταρχάς να πω ότι στηρίζω απόλυτα την άποψη του κυρίου Ντάφη για τα όσα απάντησε στην κυρία Λέζινγκ. Ακόμα και αν είμαστε πολύ ακριβείς, όταν αυτά τα πράγματα φτάνουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και τη συζήτηση μεταξύ των κρατών μελών, ε, θα είναι όλα θέμα ερμηνείας. Ακόμα και αν είναι πολύ αυστηρά τα πράγματα. Γιατί λοιπόν να μην δώσουμε περισσότερη ευελιξία γιατί ούτως ή άλλως όλα θα είναι θέμα ερμηνείας. θέμα ερμηνείας για παράδειγμα είναι να είστε κάποιες φορές υπέρ κάποιων χωρών που ε, ε, κάποιες άλλες φορές δεν θα κάνετε καν τον κόπο να ασχοληθείτε με μια επίθεση εναντίον τους ή ε, με το γεγονός ότι τους έπληξε κάποια καταστροφή. Το να επιτρέψουμε λοιπόν στις χώρες, θα πρέπει να, να επιτρέψουμε στις χώρες να βρουν το σωστό βηματισμό για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν την κατάσταση. Δεύτερον, για τα όσα λέει ο κύριος Νταφ ε, για τον τίτλο. Το άρθρο 7 λέει ότι σε περίπτωση επίθεσης κατά των κρατών μελών, αυτό λέει στην αρχή, μετά λέει ότι οι χώρες θα παρέχουν όποια μορφή συνδρομής μπορούν, ε, ουσιαστικά δηλαδή είναι επανομοιότυπο με το άρθρο 5. Ε, Όπως συζητήσαμε εδώ λοιπόν, θέλαμε να κάνουμε μια διάκριση μεταξύ μιας ρήτρα αλληλεγγύης, η οποία είναι κάτι το οποίο κατά πάσα πιθανότητα θα χρησιμοποιηθεί συχνότερα από την, την άλλη δυνατότητα, και εδώ συμφωνώ μαζί σας, ότι είναι κάτι πιο ειδικού χαρακτήρα. Αν όμως ε, ε, περάσουμε σε ψηφοφορία θα ψηφίσουμε και τελικώς θα αποφασίσουν ε, οι κάλπες. Ευχαριστώ. <laughs> Euh, Μάλιστα. Δεν υπάρχουν άλλες παρεμβάσεις. Επομένως, συνεχίζουμε. Στην ΑΦΕ τον Οκτώβριο στο Στρασβούργο θα γίνει ψηφοφορία. Και πάλι τώρα ο κύριος Πασκού όμως, ο οποίος ακατάπαυστα συνεχίζει για να μας μιλήσει για την γνωμοδότησή του, την οποία η υποεπιτροπή μας πρέπει να συντάξει, όσον αφορά τον ενωσιακό μηχανισμό πολιτικής προστασίας. γνωμοδότηση την οποία πρέπει να υποβάλουμε. Η καθήλυνα αρμόδια επιτροπή είναι η Επιτροπή Περιβάλλοντος. Η κυρία Γκαρντίνη είναι η συγγήτρια στην Επιτροπή Περιβάλλοντος. Έχουμε λοιπόν ένα σχέδιο γνωμοδότησης από τον κύριο Πασκού. Μπορείτε να υποβάλλετε τροπολογίες μέχρι τα τέλη της εβδομάδας. 12 Οκτωβρίου, 12 το μεσημέρι. Ιωάννα. Uh, ναι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας παρουσίασε σε εμά και στο Συμβούλιο μια πρόταση απόφασης για ένα ε, μηχανισμό πολιτικής προστασίας της Ένωσης, ο, ο οποίος ενισχύει νέες δυνατότητες για να προλαμβάνουμε και να απαντούμε σε καταστροφές και εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Επικράτειας. Η γενικότερη προσέγγιση μας βρίσκει σύμφωνους και θα θέλαμε τα παρόντα ad συστήματα ε, να μεταμορφωθούν σε ένα ε, μηχανισμό ε, αντιμετώπισης των καταστραφών προληπτικά, σεβόμενοι ταυτόχρονα και τις δομές πολιτικής προστασίας των κρατών μελών. Το βασικό θέμα που μας απασχολεί είναι να διασφαλίσουμε ότι έχουμε διαχείριση πρόληψης και να δημιουργήσουμε και ένα πουλ υποδομών ε, σε αναμονή, που, ε, γεγονός που σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να περιμένουμε να βρεθούμε εν μέσω κρίσης για να αντιμετωπίσουμε μια κατάσταση και να δούμε τι θα κάνουμε, αλλά να έχουμε προσχεδιασμένα κάποια πράγματα. Μία προσέγγιση προληπτική. Επίσης θα θέλαμε να αναβαθμίσουμε τον τρέχοντα μηχανισμό συντονισμού. Υπάρχει ένα κέντρο ενημέρωσης και θα πρέπει να εξοπλιστεί καλύτερα, ε, να έχουμε ένα κέντρο αντιμετώπιση καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης ε, και να λειτουργεί 24 ώρες το 24 ώρο, 7 μέρες την εβδομάδα για να μπορέσουμε να αναπληρώσουμε κενά δυνατοτήτων από ε, δυνατότητες που χρηματοδοτούνται σε επίπεδο ένωσης. Διότι υπάρχουν διάφορες περιπτώσεις ε, στις οποίες ναι μεν κάποιος έχει τις δυνατότητες να τις αντιμετωπίσει ενώ σε κάποιες άλλες περιπτώσεις μπορεί να μην έχουμε τα μέσα που χρειαζόμαστε. Επίσης να υπάρχουν δυνατότητες ε, να καλύπτονται κυρίως ε, το κόστος μεταφοράς. Ε, αυτό πρέπει να το έχουμε υπόψη, να θέλουμε να είμαστε αποτελεσματικοί και να βρισκόμαστε επί τόπου και επίσης να είμαστε κατάλληλα προετοιμασμένοι και να μπορέσουμε να βοηθήσουμε και τα εθνικά προγράμματα διαχείρισης πολιτικής προστασίας. Να ξέρουμε λοιπόν τι κάνουν οι άλλοι, να είμαστε προετοιμασμένοι και εμείς, να υπάρχει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση και να γνωρίζουμε καλύτερα τι πρέπει να κάνουμε σε αυτές τις περιπτώσεις. Προτείναμε ένα σχέδιο γνωμοδότησης, ε, ε, προτείνουμε πέντε τροπολογίες ε, κυρίως για να στηρίξουμε καλύτερη ενσωμάτωση των συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης πολιτικής προστασίας με τα υπόλοιπα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης. Θέλουμε να υπάρχει συνέπεια με τη μελλοντική εφαρμογή της ρήτρα αλληλεγγύης, την οποία συζητάμε. Θέλουμε να υπάρχει ένα σαφής σύνδεσμος μεταξύ του μηχανισμού και της ενεργοποίησης αυτής της ρήτρα αλληλεγγύης και φυσικά ε, συνεργασία με τα μέσα κοινή πολιτικής ασφάλειας και άμυνας. Τέλος, ε, δεν παρουσιάσαμε τροπολογία για το άρθρο 16, το οποίο άρθρο αναφέρεται στη σχέση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, διότι Υπάρχει ήδη συμφωνία μεταξύ Συμβουλίου και Ευρωπαϊκής Επιτροπής επί του ζητήματος αυτού και αν παρουσιάσουμε και εμείς άλλη τροπολογία, τότε θα ξεκινήσει μια ε, εντελώ νέα κατάσταση, ενώ στην πραγματικότητα αυτό που θέλουμε είναι να περάσουμε από τη συζήτηση στην απτή εφαρμογή, σε περίπτωση που το χρειαστούν φυσικά οι χώρες μέλη. Εφόσον δεν υπάρχει συμφωνία δεν υπάρχει πρόβλημα, αλλά εάν υπάρχει συμφωνία θα πρέπει να την τηρήσουμε και ε, νομίζω ότι αυτό το κατανοούν όλοι. Πρέπει να γίνεται σεβαστή συμφωνία. Αυτά λοιπόν από πλευρά μου. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να πάρει το λόγο, κύριο Στά. Μπορείτε να μας παρουσιάσετε λοιπόν πώς έχουν τα πράγματα, πώς έχει η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Thank you very much, Mr. Chairman. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλησπέρα σας. Θα ήθελα να ξεκινήσω ευχαριστώντας τον κύριο Πάσκου για τη δουλειά που έκανε. Ήμασταν σε στενή συνεννόηση και νομίζω αυτό θα φανεί στο τέλος. Να πω λίγα λόγια για να αντιληφθούμε γιατί η Κομισιόν έκανε αυτές τις προτάσεις. Υπάρχουν στατιστικά δεδομένα που δείχνουν πως υπάρχει αύξηση στον αριθμό και συχνότητα των καταστροφών και παγκοσμίω και εντός της Ένωσης. Αυξάνονται λοιπόν και ταυτόχρονα εμείς είμαστε και πιο ευάλωτοι. Όσο πιο περίπλοκες είναι οι οικονομίες και οι κοινωνίες μας, τόσο πιο ευάλωτοι είμαστε και τόσο πιο μεγάλη οικονομική ζημία. Το είδαμε αυτό στην Ιταλία όταν ένας σεισμός καταλήξει σε πάρα πολύ μεγάλες οικονομικές ζημίες για μια περιφέρεια. Αυτό είναι σημαντικό λοιπόν. Αυξάνονται οι καταστροφές και πρέπει να είμαστε έτοιμοι ταυτόχρονα και αυτό είναι το δεύτερο στοιχείο στο οποίο έρχομαι. Εδώ έχουμε με στήριξη των Ευρωπαίων πολιτών για να κάνουμε περισσότερα. Τα αποτελέσματα του Ευρωμπαρόμετρου δείχνουν πως πάνω από το 90% των πολιτών μας θέλουν πιο συντονισμένη προσέγγιση για να είμαστε προετοιμασμένοι για καταστροφές. Οι πολίτες μας θέλουν να συνεργαζόμαστε και ελπίζουμε να μπορέσουμε να ζητήσουμε και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που για πρώτη φορά θα συνομοθετεί να υλοποιήσει αυτή την έκκληση. Ο κύριος Πάσκου ανέφερε τα κύρια στοιχεία της πρότασης. Δεν χρειάζεται να μπω σε λεπτομέρειες, αλλά με λίγα λόγια. Νομίζω πως η όλη πρόταση αφορά την, την οικονομία, δηλαδή να επιτύχουμε περισσότερα με λιγότερους πόρους, αυξάνονται οι ανάγκες, μειώνονται οι δημόσιοι πόροι, οπότε υπάρχει ένα, μια ψαλίδα μεταξύ των αναγκών που προκύπτουν από τις καταστροφές και των πόρων. Οπότε η μόνη λύση είναι να γίνουμε πιο αποτελεσματικοί και να δούμε τη δυνατότητα ευρωπαϊκού συντονισμού και συνεργασίες. Και αυτό για εμάς συγκεκριμένο μεγαλύτερο βάρος στην πρόληψη, προφανώς οποιοδήποτε ευρώ ξοδεύεται σε πρόληψη σημαίνει 7 ευρώ σε θεραπεία σύμφωνα με τις μελέτες πρέπει να επενδύσουμε στις μελέτες να ξέρουμε το τι θα γίνει ποιος θα κάνει τι όταν γίνει η καταστροφή και ποιοι πόροι θα έρθουν από πού και αυτό βεβαίως σημαίνει λύσεις επιμελητίας μεταφορών και οικονομικές Συνολικά λοιπόν αυτό το οποίο προσπαθούμε να κάνουμε είναι να βρούμε μια προσέγγιση σχεδιασμού, σεβόμενη βεβαίως και την αρχή της επικουρικότητας, καθώς τα κράτη-μέλη την κυρία ευθύνη. Ο μηχανισμός είναι διαθέσιμος ε, για χρήση εντός της Ένωσης και εδώ πέρα θέλω να είμαι σαφής η πρώτη χρήση βεβαίως αφορά τις καταστροφές εντός της Ένωσης αλλά Έχουμε δει τα τελευταία χρόνια πως υπάρχει και κάποια αξία στο να προσφέρουμε αυτή τη στήριξη σε τρίτες χώρες όταν τις ε, πλήττουν καταστροφές. Όσον αφορά τώρα το σχέδιο έκθεση του κυρίου Πάσκου, μπορώ να πω πως εμείς καλωσορίζουμε τις που προτείνονται όσον αφορά τη σύνδεση με τη ρήτρα αλληλεγγύης. Είναι ξεκάθαρη πως υπάρχει αυτή η σύνδεση. Φαίνεται αυτό στο κείμενο η ανάγκη για πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση και σύνδεση με άλλα συστήματα έγκαιρης προειδοποίηση, οπωσδήποτε ενισχύει την Κομισιόν και ήδη κάνουμε πολλή δουλειά στον τομέα αυτών, όπως και η ανάγκη ανάπτυξης περαιτέρω συνεργειών. Θα μείνω σε αυτά. Εάν υπάρχουν ερωτήσεις, οπωσδήποτε είμαι στη διάθεσή σας. Ευχαριστώ. Merci Σας ευχαριστούμε. Εξ ονόματος Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης, θέλει κάποιος να πάρει το λόγο. Κύριε Πιζάνη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κοιτάξτε, δεν έχουμε να κάνουμε συγκεκριμένε παρατηρήσει. Νομίζω ότι τα πιο σημαντικά πράγματα τα είπε ήδη ο συνάδελφο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Πρόεδρο. Ευχαριστούμε πολύ. Πολύ σύντομα θα με αντικαταστήσει ο συνάδελφος Γκάλερ γιατί γίνεται ψηφοφορία στην ε, Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων για το βραβείο Ζαχάροφ. Νομίζω ότι ε, θα ήθελε να επιμείνει σε κάποια σημεία, ιδίως ε, όσον αφορά την κοινή χρήση των μέσων πολιτικής προστασίας μας λέει ουσιαστικά ότι θα ήθελε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επέμβει προκειμένου να βοηθήσει, να συντονίσει, αλλά να μην αντικαταστήσει τελικά τα κράτη-μέλη. Τα κράτη-μέλη είναι αυτά τα οποία θα πρέπει να είναι αρμόδια για την όλη διαδικασία. Και αυτό άλλωστε έχουμε πει και σε προηγούμενα ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και επίσης θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης να ελέγχει την όλη συνέπεια της δράσης Ευρωπαϊκής Ένωσης στα πλαίσια της κοινή πολιτική άμυνα και ασφάλεια. Ουσιαστικά ελέγχεται κάθε φορά ότι ακολουθούμε του στόχου που έχουμε θέσει στα πλαίσια τη κοινή πολιτική άμυνα και ασφάλεια. Ο κύριος Γκάλερ άμεσα θα, όταν επιστρέψει θα σα αναφέρει περισσότερα σχόλια ενδεχομένω. Κυρία Λέζινγκ έχει το λόγο. Äh, ναι, βεβαίως συμφωνούμε με την προσπάθεια μεγαλύτερης αποτελεσματικότητας, ε, σχεδιασμού για τις καταστροφές. Υποστηρίζουμε τις προτάσεις για καλύτερη εκπαίδευση, απόσπαση ειδικών κτλ. Δεν θεωρούμε όμως πως η στρατιωτικοπολιτική συνεργασία ή η στρατιωτικοποίηση της προστασίας από καταστροφές είναι σωστή. Οπωσδήποτε υπάρχει η πραγματικότητα. Δηλαδή, εάν δίνονται συνεχώς κονδύλια στο στρατό και όχι στην πολιτική προστασία, τότε υπάρχουν πολύ περισσότερες δυνατότητες ε, στις ένοπλες ε, δυνάμεις και άρα πάει λέγοντας. Στη Γερμανία, παραδείγματο χάρη, έχουμε και οργανώσεις ε, πολιτικής προστασίας, και ε, το λεγόμενο Technisys Hillsback που εργάζεται και στο εξωτερικό και έχει δείξει πως ε, υπάρχει δυνατότητα πολιτικής προστασίας από τις καταστροφές. Εδώ θεωρώ πως υπάρχει σοβαρός κίνδυνος για τη δημοκρατία ε, Επίση, τα περιγράφουν τελείως διαφορετικά η ΜΚΟ, με άλλες αποχρώσεις. Δηλαδή, μετά από καταστροφές, ο στρατός έρχεται βοηθάει και δεν φεύγει. Οπότε εμεί ζητάμε να υπάρξει εξοπλισμός αποτελεσματικός όλων των πολιτικών οργανισμών για να μην χρειάζεται στήριξη από το στρατό. Ευχαριστώ. Η συζήτηση αυτή έχει γίνει πολύ συχνά και μερικές φορές πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί διεξάγεται με τον τρόπο αυτό. Ιωάννη, ενδεχομένω θα ήθελες στο λόγο για να κλείσει αυτός ο πρώτος γύρος παρατηρήσεων τουλάχιστον. Να πω και εγώ τα τελευταία λόγια. Για άλλη μια φορά σας ευχαριστώ πολύ. Και σίγουρα θα πρέπει να βρούμε μια ισορροπημένη προσέγγιση. Να ανταποκριθούμε από τη μια στα αιτήματα αυτά που ακούσαμε ότι υπάρχουν όλο και περισσότερες καταστροφές και από την άλλη να ανταποκριθούμε στην όλο και διαφορετική φύση των καταστροφών αυτών. Ξέρετε ότι στην Φουκουσίμα είχαμε στην αρχή α, το σεισμό, στη συνέχεια το τσουνάμι, στη συνέχεια το πυρηνικό ατύχημα. Καταλαβαίνετε ότι στην περίπτωση αυτή έπρεπε να αντιμετωπίσουμε τρεις διαφορετικές περιπτώσεις, τρεις διαφορετικούς κινδύνους. Αυτή είναι η πραγματικότητα πλέον και πρέπει από τη μια να δούμε πώς θα καταφέρουμε να εξορροπήσουμε την παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και όλοι θα απευθυνθούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέγοντας της μα τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξέρουμε λοιπόν ότι θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε πλέον καλύτερα τα μέσα τα οποία διαθέτουμε, να γίνουμε δηλαδή πιο αποτελεσματικοί. Από την άλλη όμως τα μέσα αυτά εξακολουθούν και παραμένουν εθνικά μέσα. Ξέρετε ότι τα κράτη-μέλη θα εξακολουθούν να είναι τελικά υπεύθυνα για το τι μπορούν να παράσχουν για την επέμβαση, για την τελική μορφή που θα πάρει τελικά η επέμβαση. Επομένως, ε, ο κύριος Γκάλερ έχει δίκιο ότι θα πρέπει να διευκολύνουμε τα κράτη-μέλη για να παρέχουν τα μέσα αυτά σε ευρωπαϊκό επίπεδο, προκειμένου αυτά να καταστούν αποτελεσματικά. Για την ε, στρατικοποίηση, ε, κανείς δεν θέλει ουσιαστικά να θέσει εκτός τον ε, στρατό από τις αρμοδιότητες που έχει για την ασφάλεια και τις άμυνας μιας χώρας και να το τοποθετήσει στην δική μας την πολιτική προστασία που συζητάμε σήμερα. Η παρουσία του στρατού δικαιολογείται γιατί πολλές φορές είναι οι μόνοι που είναι παρόντες σε ένα σημείο που προκαλείται ένα ατύχημα, μια καταστροφή, είναι οι μόνοι που έχουν τον απαραίτητο εξοπλισμό και τα απαραίτητα μέσα. Τους καλούμε λοιπόν να λάβουν δράση μέχρι να κινητοποιηθούν οι υπόλοιποι μηχανισμοί πολιτικής προστασίας συμφωνώ μαζί σας ότι θα πρέπει να έχουμε καθαρούς μηχανισμούς πολιτικής προστασίας, όσο όμως δεν υφίστανται οι μηχανισμοί αυτοί, θα πρέπει να συνεχίσουμε να απευθυνόμαστε και στο στρατό. Δεν θα πρέπει να παραγωνίσουμε ενδεχομένω την βοήθεια που μπορεί να μας παρέχει ο στρατός ή την υποστήριξη την οποία παρέχει. Πρέπει κατά περίπτωση κάθε φορά να προχωράμε ρεαλιστικά. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Θα συνεχίσουμε προφανώς τη συζήτηση για το ζήτημα αυτό. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δοθεί έντονη προβολή στην κοινή γνώμη όσον αφορά το ζήτημα αυτό. Είναι πολύ σημαντική παρατήρηση αυτή και ελπίζω ότι θα καταφέρουμε να βελτιώσουμε τα συστήματα αυτά ανταπόκρισης ε, προστασίας. Πολλές φορές δίνει την εντύπωση ότι ακόμα και οι αποτελεσματικές παρεμβάσεις τελικά παραμένουν αρκετά κατακαιρματισμένες και δεν έχουν την απαραίτητη προβολή σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Επομένω και, το, και η πτυχή αυτή είναι πολύ σημαντική. Πολύ ωραία. Ολοκληρώνεται η εξέταση αυτής τη γνωμοδότηση για σήμερα. Και θα συνεχίσουμε με την συνεδρία του Προεδρείου. Σας ευχαριστώ πολύ. Euh, Πέντε 5 5 λεπτά διάλειμμα. 3, 3 λεπτά διάλειμμα.